Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος βουλευτής Μάρκος Φέμπερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να ακούσετε, αν δεν θέλετε να ακούσετε τον κύριο Φέρμπερ, σκανδαλώδες, λέει ο κύριο Φέρμπερ, σας παρακαλώ να εξέλθετε τις θέσεις Κυρία Χάρμψη, για παράδειγμα. Κυρία Χάρμψη, καλά θα κάνετε να με ακούσατε πριν βγείτε στι ε, τύπου αύριο. Καθίστε παρακαλώ. So, bitte sehr, Herr Kollege. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για πρώτη φορά σήμερα συζητάμε συγκεκριμένη νομοθεσία μετά την υπόθεση LuxLeaks. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση, γιατί το θέμα είναι ως Κοινοβούλιο να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για διαφάνεια, σαφήνεια, δίκαιη φορολογική φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ιδιαίτερα στο θέμα της φορολογίας τα κράτη-μέλη υποχρεούνται ήδη σήμερα να ανταλλάσσουν πληροφορίες, αλλά έως τώρα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει, για να το πω ευγενικά. Θα ήθελα λοιπόν ευθύ εξ αρχή να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επίτροπο Ανταγωνιστικότητας που προωθεί το θέμα της δίκαιης φορολόγησης και στο πλαίσιο των κρατικών επιδοτήσεων, γιατί δεν είναι τίποτα διαφορετικό στην τελική ανάλυση ο άδικο φορολογικό ανταγωνισμό. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή τη. προκειμένου όλοι οι φορολογικοί συντελέστέ διασυνοριακά να μπορούν να ενταχθούν σε μια αυτόματη διαδικασία. Και θεωρούμε ότι η πρώτη αυτή προσέγγιση είναι καλή, αλλά στην Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων ε, η πρότασή μας περιλαμβάνει πολύ πιο πολλά μέτρα και θα ήθελα να αναφέρω κάποια ενδεικτικά. Ο τομέας εφαρμογής. Είπαμε με σαφήνεια ότι θα θέλει... Σας παρακαλώ κύριε Μπρόκ, είτε βγείτε είτε καθίστε. Κύριε Μπρόκ, σας παρακαλώ. Βγείτε έξω, μην κάνετε φασαρία. Είπαμε λοιπόν στον τομέα εφαρμογής όλες οι φορολογικές αποφάσεις ε, όσο δεν αφορούν ε, φυσικά άτομα αλλά νομικά πρόσωπα να συμπεριληφθούν σε αυτή τη διαδικασία. Για νομικά λοιπόν πρόσωπα, για όλα τα νομικά πρόσωπα, σαφής ε, διαβρύνση. Επίσης είπαμε να υπάρχει άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, όχι κάθε τρεις μήνες όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ε, ζητήσαμε επιπρόσθετες ε, πληροφορίες να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο αυτό. Ένας ε, φορολογικός, αριθμός φορολογικού μητρώου, παραεκκλήσεις από το κανονικό φορολογικό δίκαιο και το καθεξής. Και είπαμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στα πλαίσια του δικαίου του διαγωνισμού να εφαρμόζει τις αποφάσεις αυτές. Για τόσο σημαντικό σημείο γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε να υπάρχει ένα φορολογικό δίκαιο το οποίο δεν θα στρέφεται κατά των γειτονικών χωρών, αλλά να ξέρει κανείς ότι οποιαδήποτε φορολογική απόφαση θα πρέπει να λάβει υπόψη και τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, κανόνες για τις επιδοτήσεις. Και είμαι απογοητευμένος για το γεγονός ότι το Συμβούλιο στις 6 Οκτωβρίου συμφώνησε επί μιας ε, συμφωνίας η οποία είναι πολύ κατώτερη αυτών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο τη συνοριακή δηλαδή ε, απόφαση, τη συνοριακή φορολογικές αποφάσεις, ε, χωρίς όμως να ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνεται. Είναι ασαφές το Συμβούλιο. Η θέση σε ισχύ να παραταθεί κατά ένα έτος με αναδρομικό χαρακτήρα πέντε ετών και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι είμαι απογοητευμένος. Και πολύ λυπάμαι που οι υπουργοί του Συμβουλίου δεν έλαβαν υπόψη και δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της Επιτροπής μας. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση προς τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν σοβαρέ διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το θέμα τη φοροδιαφυγή προαποφύγη, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σαφέ ευρωπαϊκό διαφανέ μοντέλο που δεν θα επιτρέπει να υπάρχουν φορολογικά συστήματα ει βάρον των γειτονικών χωρών και να φορολογείται το κέρδος εκεί που δημιουργείται και χαίρομαι για το γεγονό ότι καταφέραμε να πετύχουμε ευρεία συνένεση στην Επιτροπή. Ελπίζω το ίδιο να συμβεί και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η, κυρία Φερέιρα που αντικαθιστά τον κύριο Κόφουτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Κύριε Επίτροπε, μα τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Και είπα κάτι, είπα. μα. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Πρόεδρε να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του και την Επιτροπή μας που συλλογικά εργάστηκε για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Αγόρτερα σήμερα το βράδυ στην Ειδική Επιτροπή Τάξη που δημιουργήθηκε μετά από το σκάνδαλο LuxLeaks θα εξετάσουμε άλλη έκθεση και ελπίζουμε πως το πνεύμα συνεργασίας θα κυριαρχήσει. Πέρασε ένας ε, χρόνος από τη ε, σκάνδαλο του Λουξ Λίξη και το πρόβλημα ανταλλαγή πληροφοριών εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να εξεταστεί κατεπηγόντως και σοβαρά μέσω συμβιβαστικών λύσεων, όχι μόνο εντός του Κοινοβουλίου, αλλά και μέσω μιας διαθεσμικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο με τρόπο ώστε να εισαχθεί μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ένας νέος τρόπος για να ε, προσεγγίσουμε προσεγγίζουμε τα θέματα τα φορολογικά. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντα την Κομισιόν για την πολυάριθμε πρωτοβουλίε που ήδη έφερε προ συζήτηση και να τη ζητήσω να μην σταματήσει αυτόν τον αγώνα και αυτή την προσπάθεια. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια στεναρή στάση αυτού του Κοινοβουλίου που προσπαθούμε να την οικοδομήσουμε. Είναι απαραίτητο μια, να έχει μια ισχυρή θέση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και μια αξιόπιστη θέση οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει από του Συμβουλίου. Προ αυτή την κατεύθυνση συγκλίνω με τα όσα μόλι έλεγε ο συνάδελφο Φέρμπερ σε σχέση με τις την, την απογοήτευση που μας προκάλεσαν οι αποφάσεις της 6ης Οκτωβρίου του ΕΚΟΦΗΝ. Όχι μόνο λόγω της έναρξης ισχύω των νέων διαδικασιών, αλλά και για τρία σε άλλου λόγου. Καταρχήν, είναι απαράδεκτο η Συμφωνία Ανταλλαγή Πληροφοριών, συμφωνίε που ήταν μέχρι τώρα μυστικέ και που ευνοούσαν τις πολυεθνικές σε θέματα φορολογία, να ε, προσαρμόζονται και να συνάπτονται ε, μεταξύ των κρατών μελών χωρίς να αποδίδεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ρόλος τον οποίο πρέπει να παίξει, που πρέπει να είναι δηλαδή η βάση για αυτή την ανταλλαγή των πληροφοριών, έτσι ώστε να αποφεύγεται γίνεται αυτό που αποτέλεσε την διάλυση όλων των διακρατικών συμφωνιών ανάμεσα στα... και που συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι τώρα να συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι η βάση ανταλλαγή ε, αυτών των συμφωνιών. Επίση θα πρέπει αυτή η ανταλλαγή ε, πληροφοριών ε, να πάψει με αυτέ τι αποφάσει ειδική ευνοϊκή εφορολογική μεταχείριση. Όταν δηλαδή εξακολουθούσαν να ισχύουν οι προηγούμενες οδηγίες και άρα να ελεγχθούν όλες οι συμφωνίες οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ανάμεσα στα κράτη για αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ήθελα εξίσου να αναφερθώ στο γεγονός ότι όλα τα rulings, οι ειδικέ αυτές συμφωνίες ε, για ευνοϊκή φορολογία να διαβιβάζονται στην Κομισιόν. Γιατί στην εσωτερική αγορά τα πλεονεκτήματα που δίνονται από ένα μόνο κράτος μέλος σε μια πολυεθνική εταιρεία έχουν αυτόματα αντίκτυπο και στις υπόλοιπε. Ε, χώρες. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα να περιορίζεται η υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών μόνο στις συμφωνίες που γίνονται ανάμεσα σε κράτη. Από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία, το ruling, δημιουργεί Μία πρόβλημα στην ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά δημιουργεί, προκαλεί κίνδυνο απώλειας φορολογικής για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ε, θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια προβλημα στην ευρωπαικη στην ευρωπαικη ατζέντα για αυτά τα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται από αυτού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται τατικά, όμως το Συμβούλιο θα πρέπει να δράσει με ρεαλισμό, αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να διορθωθεί αυτή η κατάσταση ε, φορολογικής αδικίας στην Ευρώπη και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των Ευρωπαίων πολιτών που είναι αυτοί που καταβάλουν τους φόρους στο κάτω-κάτω. Να αποκατασταθεί λοιπόν η αξιοπιστία στην εργασία σε αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, σχέδιο, στο οποίο όλοι μας θέλουμε να πιστεύουμε. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα έχει το λόγο ε, ο τρίτος εισηγητής που είναι η κυρία Σκοτ Κάτω. Εμείς βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις δεν προσανατολίζονται μόνο σε τοπικά νησιά αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν με τις ε, πολυεθνικές. Οι πολίτες πλέον το τίμημα. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάνουν και οι επενδύσεις αποδυναμώνονται. Οι πολυεθνικές μπορούν να ρυθμίσουν τα πρώτα θέματα ευκολότερα. Η φορολογία και η φορολογική δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά σημαντική για τους πολίτες της Ένωσης προσεγγίζουμε την επέτειο του σκάνδαλου των LuxLinks, θέλω να σταθώ σε ένα βασικό θέμα της συζήτησης αυτού. Το ποιος πρέπει να ξέρει τι για τα φορολογικά. Τι ξέρουμε. Η απάντηση είναι ότι ξέρουμε πολύ λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να ξέρουμε για να διαμορφώσουμε πολιτικές που θα διασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, ότι οι επιχειρήσεις πληρώνουν αυτά που οφείλουν. Ω ερετή εκπρόσωπο και μέλο τη Επιτροπή Τάξε, πολλά κείμενα παραμένουν στα οποία δεν είχα πρόσβαση. Τον περασμένο Νοέμβριο όλος ο κόσμος στην Ευρώπη με τρόμο διαπίστωση ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής ήταν αρχιτέκτονας ενός συστήματος για την διευκόλυνση, τη φορική διευκόλυνση των μεγάλων επιχειρήσεων. Χωρίς τον Αντώντελ Τούρ και τις θαραλές δράσεις του δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτά. Πώς είναι σωστό λοιπόν ο Ντελτούρ να διώκεται αυτή τη στιγμή ενώ οι αρχιτέκτονες αυτών των ύποπτων συμφωνιών δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πολύ λίγοι από αυτούς που εκπροσωπώ πιστεύουν ότι ο ένοχος είναι ο Ντελτούρ στο θέμα της φοροαποφυγής. Το πρώτο μήνυμα ότι η Επιτροπή θέλει να πετύχει κάτι ήρθε την περασμένη εβδομάδα μετά την αναγγελία των αποτελεσμάτων για την υπόθεση των Starbucks και την ζήτηση ανάκτησης και το έτοιμο ανάκτησης πόρων. Παραμένει μακρύ ο δρόμο ακόμα. Συγχαίρω την Επιτροπή για τι δραστηριότητε τη, αλλά θα τη πρότεινα να διευρύνει τι ερευνέ τη. Φέτος το Μάρτιο η Επιτροπή υπέβαλε ένα πακέτο διαφάνειας φορολογικής που περιλαμβάνει και ένα από τα κείμενα που συζητούμε σήμερα. Προτείνουν την κατάργηση της οδηγίας του 2003 που επιτρέπει στις αρχές να, να έχουν τις πληροφορίες που θέλουν για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρξει φοροαποφυγή, αλλά που ξεπεράστηκε από, από τα νέα νομοθετικά κείμενα. Εγώ ήμουν συγκήτρια και προσπαθώ να διευκολύνω ότι δεν θα υπάρξουν παραθυράκια. Θέλω να σε ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις ε, για την υποστήριξη που έδωσαν. Η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία διαβρύνεται τώρα και ζητά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές αποφάσεις. Το κομμάτι αυτό ήταν τόσο σημαντικό που το Συμβούλιο προχώρησε και κατά παράβαση της παραδοσής χωρίς να ακούσει τη θέση της Επιτροπής και αυτό είναι κρίμα διότι εμεί βελτιώσουμε σημαντικά την πρόταση της Επιτροπής ιδίω ε, σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των στοιχείων αυτών. Επανέρχομαι στο, στο κεντρικό μου θέμα. Δεν πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο ήταν επαρκώς ε, φιλόδοξο. Ως πράσινοι ζητούμε να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις της Επιτροπής όχι μόνο για τα άλλα κράτη και την Επιτροπή αλλά και για τους πολίτες. Το αίτημα δημόσιας ενημέρωσης θα επανέλθει ως τροπολογία στην Ολομέλη διότι πιστεύουμε ότι αυτό είναι που θέλουν να μάθουν οι πολίτες της Ευρώπης. Είπα στο ξεκίνημα της ομιλίας μου το κεντρικό ζήτημα των LuxLeaks ήταν έλλειψη ενημέρωσης πολιτικοί, λογιστές, επιχειρηματίες, διευθυντές των μεγάλων επιχειρήσεων ήξεραν πολύ καλά τι εννοούν με τον όρο tax rulings. Εγώ ως βουλευτής δεν ήξερα τίποτα. Οι ψηφοφόροι μου επίσης δεν ήξεραν τίποτα. Γι' αυτό οι πράσινοι στο κοινοβούλιο το μόνο που ζητούν είναι πλήρη ενημέρωση των φορολογικών πληροφοριών. Μόνο όταν οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι οι συμφωνίε του με τι επιχειρήσει θα γίνουν γνωστέ στου ψηφοφόρου του, θα δράσουν προ όφελο των ψηφοφόρων του. Και μόνο όταν οι, οι δικηγόροι γνωρίζουν ότι θα του διώξουν, θα σταματήσουν να διαμορφώνουν νέου τρόπου φοροαποφυγή. Υπάρχει μία μπλε κάρτα. Δέχεστε να απαντήσετε. Κύριε Σκοτ, κάτω. Θέλετε να, απαντήσετε στην πράσινη κάρτα. Η κυρία Τζάνι. ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να θέσω το ερώτημα αυτό. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε οποιοδήποτε εσύ για το θέμα αυτό και εγώ πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι να ενημερώνεται σωστά το κοινό. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποιο είναι το ετήσιο φορολογικό ποσό το οποίο γλιτώνουν οι επιχειρήσεις. Ποια είναι λοιπόν η ζημιά που προκαλείται στη ευρωπαϊκή οικονομία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια αριθμητικά στοιχεία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μεγάλη και περίπλοκη ερώτηση. Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Και δεν μπορεί να θέσετε μπλε κάρτα στην Επιτροπή που έχει όμω τι πληροφορίε αυτέ. Απλώ είναι δύσκολο να κάνουμε εκτιμήσει γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία. Ένα λοιπόν από το έτοιμά σα, από το έτοιμά μας για τη δημοσίευση των φορολογικών αποφάσεων είναι για να μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο θα, τι ποσά ε, έχουν φοροαποφευθεί σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε περαιτέρω έρευνε για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του μεγέθους της κατάστασης και της απώλεια εσόδων για τα κράτη-μέλη. Ο κύριος Μοσκοβισή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνεισηγητές, η επιθετική φορολογική πολιτική είναι θέμα που ανησυχεί ιδιαίτερα την Ένωση και τον κόσμο, ιδίως στα πλαίσια των εργασιών του ΩΣΑ και της ομάδας των 20. Η αύξηση της διαφάνειας ε, στις, ε, στη φοροαποφυγή μεταξύ κρατών μελών και κομισιών είναι σημαντική φάση, σημαντικό στάδιο για την καταπολέμηση αυτής της επιθετικής ε, ε, φορολογική ε, πολιτική και τη φοροποφυγής. Αυτό είναι και το αντικείμενο των αποφάσεων τη Επιτροπή την περασμένη ε, εβδομάδα στα πλαίσια τη Fiat στο Λουξεμβούργο και του Starbucks στην Ολλανδία. Η συνεργασία μου με την κυρία Ντεστέγκερ και τι υπηρεσίε τη στο πλαίσιο αυτό είναι εξαιρετική. Σήμερα τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλο περιθώριο χειρισμού για να αποφασίσουν αν μια απόφαση φορολογικού χαρακτήρα μπορεί να έχει σημασία, να είναι ενδιαφέρουσε για άλλο κράτο μέλο της Ένωση. αυτό που αποκαλούμε ε, ανταλλαγή πληροφοριών μετά από αίτημα. Αυτό το, αυτή η έλλειψη διαφάνειας γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση από κάποιες επιχειρήσεις ε, και για τους συμπολίτε που κλήθηκαν να συμβάλλουν για τη μείωση των ελλημάτων και των, του, λόγω της κρίσης έχει γίνει κάτι το απαράδεκτο. Γι' αυτό το λόγο υποβάλαμε τον ε, Μάρτιο του 2015 μια φιλόδοξη πρόταση για την ε, δημιουργία αυτόματης ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικών καθεστώτων μεταξύ όλων των κρατών μελών. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμπερ για την ποιότητα τη έκθεσή του για την πρόταση αυτή. Είχαμε πάντα καρποφόρες συζητήσεις ε, για το θέμα αυτό. Στις 6 Οκτωβρίου τα κράτη-μέλη έφτασαν σε μια πολιτική συμφωνία που θεωρώ πολύ σημαντική δεδομένου ότι την προηγούμενη μέρα δημοσιεύθηκαν οι συστάσεις BEPS ε ε, από τον ΟΣΑ που κατόπιν εγκρίθηκαν και από την ομάδα των 20 στα πλαίσια της συνάντησης του Δέλτα Νιτάφ. Συμφωνώ με τον κύριο Λαμασούρ που προεδρεύει κόμμα της ε, Ειδικής Επιτροπής ΤΑΞ ότι οι εργασίες του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό άσκησαν σημαντικό ρόλο και μεγάλη πίεση, αποφασίστηκε πίεση προς όλα τα κρατημέλη και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Το Κοινοβούλιο δεν ήταν βέβαια στο ΕΚΟΦΗΝ. Το πνεύμα ωστόσο των εργασιών του Κοινοβουλίου βάρινε στην απόφαση αυτή. Η πολιτική αυτή απόφαση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ισχυρό μήνυμα από πλευράς της Ένωσης που μας επέτρεψε να υποβάλουμε στην Λίμα ένα κοινό φιλόδοξο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και στα πλαίσια της συνάντησης της ομάδας των 20 παρουσίασε την πρωτοβουλία αυτή ζητώντας να γίνει ένα παγκόσμιο στάνταρ. Ο κύριος Φέρμπερ εξέφρασε μια απογοήτευση και το ίδιο και η κυρία Φερέιρα. Να απαντήσω λοιπόν. Προφανώς θέσατε τρία βασικά θέματα. Ένα, τη βούληση να προχωρήσουμε παραπέρα από τις διασυνοριακές ανταλλαγές πληροφοριών, να πάρουμε όλες τις φορολογικές αποφάσεις. Μετά, έκφραση λύπης διότι ήταν μεγαλύτερη η αναδρομικότητα. Και τρίτον, ε, μια διαφοροποίηση ως προς το ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει ταχύτερα στην υλοποίηση του κειμένου. Όλα αυτά, πώς να το πω, δεν είναι ότι διαφωνούμε κύριοι και κυρίες εισηγητές. Η αρχική πρόταση της Επιτροπή άλλωστε πήγαινε πιο πέρα από αυτό που έγινε δεκτό εν τέλει στο Συμβούλιο. Κυρίε και κύριοι βουλευτές ωστόσο γνωρίζετε πώ λειτουργεί το Συμβούλιο. Πρέπει να μπορούμε να εγκρίνουμε αποφάσεις φορολογικού χαρακτήρα με ομοφωνία. Εμείς αποφασίσαμε όχι ομόφωνα αλλά και πολύ γρήγορα. Επτά μήνες μόνο χρειάστηκαν μεταξύ της υποβολής της πρώτης επιτροπής και της έγκρισης του κειμένου από το Συμβούλιο Κοφίν. Η Επιτροπή ΕΠΕΤ συνένεσε στην, ε, στο συμβιβασμό αυτό διότι η εντύπωσή μας είναι ότι οι βασικές αρχές των, το, της προτάσεώς μας περιλαμβάνονται στο κείμενο. Η ανταλλαγή των προλογικών ε, πληροφοριών αυτόματα. Το γεγονός ότι η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται μεταξύ όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, και αυτό συζητήθηκε μακρόν, η εφαρμογή από την Επιτροπή. Υπάρχει βαθμό αναδρομικότητα. Δέκα χρόνια θα ήταν καλύτερα από πέντε κατά την άποψή μου, αλλά και τα πέντε είναι καλύτερα, ταυτολογία είναι αυτό, από τα τρία για παράδειγμα που θα άρχισε να δημιουργεί προβλήματα. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση τώρα. Είχατε εκφράσει την επιθυμία να είχε ξεκινήσει ήδη στο πρώτο τρίμηνο, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016. Τα κράτη ωστόσο τόνισαν και δεν είναι παράλογο ότι ε, χρειάζεται να υπάρξει μια προθεσμία ενσωμάτωσης. Τελικά το κείμενο θα έλεγα ότι είναι αρκετά φιλόδοξο και δεν οδηγεί, και αυτό είναι ουσιαστικό κατά την άποψή μου, Αλλιώ δεν θα είχε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο η Επιτροπή, δεν αλλοιώνει την πρόταση. Είναι ένα συμβιβασμό καλή ποιότητα ωστόσο που αποτελεί, μια, αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο. Θα ήθελα να είχε παραμείνει στο κείμενο του συμβιβασμού ολόκληρο το κείμενο της Επιτροπής, αλλά θεωρώ ότι αυτό αποτελεί, είναι κάτι θετικό και για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο. Η εφαρμογή αυτή είναι σημαντική την παρακολούθηση της οδηγίας και για την ε, ε, παρακολούθηση των, της υλοποίησης από πλευράς κρατών μελών. Αν παραμέναμε μόνο σε ανταλλαγή πληροφοριών μόνο μεταξύ κρατών μελών χωρίς εμπλοκή της Επιτροπής υπήρχε κίνδυνος ε, να μην ε, πώς το πει κανείς, να τα βολεύουν μεταξύ τους οι διάφορες διοικήσεις απομακρυνόμενες από το στόχο της οδηγίας. Να πω δύο λόγια για τις άλλες δύο εκθέσεις. Πρώτον, την συμφωνία που υπογράφηκε στις 27 Μαΐου μεταξύ Ένωσης Ελβεσίας για την αυτόματη αλλαγή πληροφοριών ε, περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Αυτό είναι ιστορική σημασία συμφωνία που είναι εξαιρετικά σημαντική για τους συμβολικά διότι στην ουσία λίγοι πάβει το τραπεζικό απόρριτο της Ελβετίας για τους πολίτες. Ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση όλων των συμπολιτών μας. Και που η ανάλυση αυτή με βρίσκει σύμφωνο και τον κύριο Κοφόντ στο σχέδιο ε, ψηφίσματος και ζητώ από το κοινοβούλιο σας να ακολουθεί την άποψη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής υποστηρίζοντας την πρωτοβούλια αυτή. Επίσης, καταργήσαμε, προτείναμε την κατάργηση της ε, οδηγίας για τις αποταμιεύσεις λόγω της ε, θέσης ε, ισχύει από τον Ιανουάριο της οδηγίας που υιοθετήθηκε στα τέλη του 2014 για την αυτόματη ανταλλαγή ε, χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Είχα μια εμπειρία σε χρηματοοικονομικά στο παρελθόν και πρέπει να σας πω ότι η οδηγία για τις αποταμιεύσεις είχε, καθο... είχε υιοθετηθεί τόσο αργά που έγινε αναχρονιστική μόλις εγκρίθηκε. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με αποφασιστικό και γρήγορο τρόπο. Και τα νέα πρότυπα ξεπερνούν αυτό που θα μπορούσε να προσφέρει η οδηγία για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Χαίρομαι λοιπόν για το περιεχόμενο της έκθεσης κ. Σκότκα, το που ευχαριστώ επίσης που προτείνει την κατάργηση της οδηγίας αυτής. Μια μικρή παρατήρηση, αν μπορώ να τη κάνω. Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε για τον πρόεδρο της Επιτροπής, ε, κ. Γιούνκερ, είναι κάπως ε, ε, ε, ε αγενής. Είμαι βέβαιος ότι όταν μιλούμε για, έναν, για τον πρόεδρο ενός τόσο σημαντικού οργάνου θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε πιο σωστή φρασιολογία. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη την έκθεση για να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που υποβάλαμε για τη λειτουργία των, της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών βάσει των πληροφοριών που θέτει η οδηγία για την διοικητική συνεργασία. Στο φορολογικό τομέα, ωστόσο, εν τω μεταξύ, η Επιτροπή σίγουρα θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που έχει με τον διαρθωμένο διάλογο με την Επιτροπή, με το Κοινοβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή για να ενημερώσει ταχύτατα και αμελητή το Κοινοβούλιο για κάθε εξέλιξη. Συνοπτικά πιστεύω ότι σήμερα συζητούμε μια μίζωνα καινοτόμο αλλαγή, την επανάσταση της διαφάνειας την αποκαλώ εγώ. Ε, υπάρχουν, υπάρχει πίεση του κοινή γνώμης, η εξέλιξη των μέσων, ε, το αίτημα από πλευρά σα, το γεγονό ότι και τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευθεί πλέον να αναλάβουν δράση, όλα αυτά με πείθουν ότι με μια κοινή δράση και με τη βοήθεια των εισηγητών και βουλευτών θα προχωρήσει αυτή η επανάσταση της διαφάνειας γιατί υπάρχει πολιτική βούληση και από την Επιτροπή και από μένα ούτως ώστε κατά τα πέντε έτη της θητείας της Επιτροπής αυτής να συνεχίσουμε να προχωρούμε με αποφασιστικό τρόπο στο πλαίσιο της, ε, αποδοτής ε, πραγματικής φορολόγησης, φορολόγηση δηλαδή των κερδών εκεί που πραγματικά ε, δημιουργούνται, το τάξη, το CCTB που έχουν ε, νομοθετικά κείμενα που συμβάλλουν ε, στην φορολογική δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα κείμενα είναι κείμενα στο οποίο η Επιτροπή προχωρά και αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι σήμερα η σημερινή μέρα είναι μια, ένα στάδιο στην επανάσταση της διαφάνειας που θα συνεχίσουμε. Σα ευχαριστώ. Επόμενο ο μελετής ο κύριος Σβάμπ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι το θέμα το οποίο συζητάμε εδώ σήμερα όχι μόνο σε ό,τι αφορά το θέμα τη έκθεση του κυρίου Φέρμπερ, τον οποίο και ευχαριστώ και συγχαίρω για την εξαιρετική του εργασία, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ε, συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτα κράτη. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο λοιπόν και πολύ σύμφωνο το θέμα αυτό και θα πρέπει να προσέξουμε η βασική λογική της συνεργασίας ε, στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ε, εσωτερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπονομευτεί. Πολλέ είναι οι λεπτομέρειες τις οποίες συζητάμε εδώ. Δεν είναι καθοριστικές όμως αυτές. Αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι για τους εργαζόμενους και για τις ε, ιδιώτες θα πρέπει παρά να παραμείνει η ευρωπαϊκή ιστορική αγορά αυτό που τους υπόχαμε υποσχεθεί εδώ και χρόνια. Ένα καταφύγιο. Ύστερα, η υποχρέωση χώρα ανά χώρα δεν θα πρέπει να μπει στην λογική του 93 και να υποχρεώνουμε τις ε, επιχειρήσεις να παίρνουν πιο στα σοβαρά τις εθνικές νομοθεσίες και όχι τόσο πολύ την ευρωπαϊκή νομοθεσία παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται και απαιτήσαμε μάλιστα στην υπόθεση του Λουξλικ σε άμεση παρέμβαση και γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε και με την έκθεση ε, του κυρίου Φέρμπερ για την ε, σαφή και γρήγορη πρόθεση του συστήματος των φορολογικών ελαφρύνσεων. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσον η δυσνοριακή σημασία τέτοιων ρούλεξ, τέτοιων αποφάσεων μπορούν, μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά στα, θέμα, στα χέρια των ε, κρατών μελών ή μήπως ε, αυτό από μόνο του θα αποσταθεροποιήσει το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε σας ζητώ να συνεχίσετε τη διαδικασία αυτή που ξεκίνησε με την έκθεση αυτή και είμαστε στην αρχή της διαδικασίας και φυσικά θα πρέπει να κοιτάξουμε και την Ελβετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Σίμων. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η απόφαση κατά τη Starbucks και της Fiat της προηγούμενης εβδομάδας δεν καταδεικνύει τίποτα άλλο παρά μια καμπή στο χρόνο, γιατί έως τώρα ακούγαμε τόσο πολύ ότι η, συμπεριφορά ήταν με έναν αλλά όχι παράνομη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε στην απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας ότι μιλάμε για παράνομη συμπεριφορά κρατών και επιχειρήσεων. Και αν λοιπόν τα κράτη-μέλη όντω αυτά που ευαγγελίζονται και τις διαφορές που ζητούν ε, για το tax rulings, ε, για τις προλογικές αυτές αποφάσεις, ε, τις εννοούν στα αλήθεια για πιο πολύ διαφάνεια, πιο πολύ δικαιοσύνη, τότε μας προκαλεί εντύπωση για την τρεσή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ επιτυχή στην στο θέμα των κρατικών επιδοτήσεων γιατί μπόρεσε να δράσει βάσει του δικαίου. Αν τα κράτη-μέλη τώρα αποτρέψουν την πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ότι σκόπιμα αποφεύγουν την ε, πιο αυστηρή διαμόρφωση των κανόνων. Και γιατί, αναρωτιόμαστε, το ίδιο αφορά και τον ανδρομικό χαρακτήρα των ε, φορολογικών αυτών αποφάσεων. Αν κοιτάξουμε πότε έχουν ισχύσει αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Πρόκειται για περιόδους που καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα πέντε έτη τα οποία θα πρέπει να χορηγηθούν ως, πληροφορι... ως πληροφορίες. Άρα μήπως χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πλήρη ανταλλαγή από ε, πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά προηγούμενες ε, Πιστεύω ότι χωρί τη διαφάνεια, χωρί την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών, ποτέ στην Ευρώπη δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τι πρακτικέ αυτέ. Και ω εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, να είστε σίγουροι σίγουρος ότι μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούνα, είναι η επόμενη Ο κύριος. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η αποφυγή και η καταπολέμησή τους είναι σημαντικά ζητήματα αυτά τα οποία ε, όλους μας απασχολούν για να υπάρχει δίκαιη κατανομή του φορολογικού άχθου. Συζητάμε δύο τεχνικά ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένα και θα προσαρμόσουν την νομοθεσία μας σε διεθνή πρότυπα και αυτά είναι πολύ θετικά και συζητάμε και ένα τρίτο θέμα το θέμα τη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για το tax rulings για τι φορολογικές ελαφρύνσεις. Και εδώ έχω κάποιε ερωτήσει να θέσω. Ήμουν πολύ ικανοποιημένο με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά είναι ουσιώδη. Και ο Γιώχαν Φανάμφερφελτ, ο Υπουργό Οικονομία μα, θα ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου να διαβιβάζει τι πληροφορίε αυτέ στα άλλα κρατημέλια, αλλά μετά πέρασε στο Κοινοβούλιο από την Επιτροπή το θέμα αυτό και εδώ πέρα νομίζω ότι στράβωσαν κάποια πράγματα και σε κάποια... Σε κάποια τροπολογία στο Κοινοβούλιο φαίνεται ότι υποστηρίζει την ε, γραφειοκρατία και τις σκοτεινές διαδικασίε. Αυτό λοιπόν δεν το χρειαζόμαστε. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα πιο αποτελεσματικά μέσα, στα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και Θεωρώ ότι αυτό είναι το διακύβευμα με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Για ένα παράδειγμα να σας δώσω. Γιατί να ανταλλάσσουμε όλα τα tax ruling σε όλες τις φορολογικές ελαφρύνσεις και να μην κοιτάμε μόνο τις φορολογικές αυτές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με διασυνοριακό χαρακτήρα. Πίστευω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε λάβει καλύτερες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. σε ja σας ευχαριστώ. Γεζικ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, δεν θέλουμε να ε, παρέμβουμε στις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Ωστόσο θα έπρεπε να είναι παράνομες οι φορολογικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε κάθε μεγάλες εταιρείες να ωφελούνται σε κάποιες χώρες. Ε, αυτές, αυτά τα tax rulings διευκολύνουν επιχειρήσεις για να αποφύγουν να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο τους σε φόρους, αλλά διευκολύνουν και κράτη-μέλη, ε, γιατί αυτά έχουν τα, την ευθύνη όσον αφορά τη δίκαιη φορολογία. Αυτή η έρευνα αποδεικνύει ακόμη μια φορά πως είναι πολύ σημαντικό να δίδεται στην Κομισιόν ο κεντρικός ρόλος ε, στη διαδικασία της αυτόματης ανταλλαγής των πληροφοριών, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον κοινοτικό νόμο. Ελπίζω πως τα κρατημέλη θα αποκομίσουν τα διδάγματα αυτών των υποθέσεων και θα συμφωνήσουν να δώσουν πρόσβαση στα έγγραφα στην Κομισιόν, να εξασφαλίσουν ότι τα, οι ευρωπαϊκές εταιρείε ε, αντιμετωπίζονται επίσης όρις. Το κείμενο της έκθεσής μας πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και ζητά τι ισορροπημένες ε, διατάξεις για τη διαφάνεια. Κατανοώ ότι ορισμένοι θα θέλαν πλήρη πρόσβαση σε αυτές τις αποφάσεις, στις φορολογικές ρυθμίσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να δίνονται αυτές οι πληροφορίες στην Κομισιόν. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους κοιόδης για την εργασία τους ε, που κατέληξε σε καλή έκθεση. Ε, κατά τη γνώμη μου, με, με σχετικά περιορισμένο αριθμό τροπολογιών που θα πρέπει να ψηφιστούν και είμαι ευτυχής που πάει ενάντια στο ρεύμα που συχνά ψηφίζουμε κατά τμήματα για κάθε κόμμα και τελεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Ματίας Μαρίζα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου οι 19 από τις 20 εταιρείε που ε, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο πληρώνουν τους φόρους τους σε άλλες χώρες όπου δημιουργείται μια, ένας αγώνας ε, για την εγκατάσταση των εταιριών εκεί όπου ε, είναι χαμηλότερη η φορολογία. Αυτή η, η νομοθεσία την οποία συζητάμε εδώ δεν θα επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το φαινόμενο. Να εξασφαλίσουμε την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ε, φορολογικές αρχές είναι ε, μια βασική δικαιοσύνη και γι' αυτό συγχαίρω τον κύριο Φέρμπερ έχουμε φόρους που διαφεύγουν και που υπολογίζονται σε 50 με 70 ε, δις ευρώ. Εάν υπολογίσουμε και ένα ποσό που σχετίζεται με την φοροδιαφυγή και τις ειδικέ συμφωνίες, αυτά τα ποσά μπορεί να ανέρχουν σε 170-190 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η απάτη λοιπόν επιβαρύνει τους φορούς που επιβάλλονται στους εργαζόμενους και στους υπόλοιπους φορολογούμενους ε, ενώ ταυτόχρονα στερούν από τα κυρίαρχα κράτη βασικούς πόρους για να μπορέσουν να ασκήσουν την κοινωνική τους πολιτική, να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα και για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Για όλα αυτά η οικονομική και η κοινωνική ανισότητα αυξάνονται λόγω όλων αυτών. Μια βασική δράση για την ε, διαφάνεια είναι αυτή η συμφωνία. Ε, γι' αυτό και καλό του συναδέλφους να στηρίξουν τις τροπολογίες που βάλουμε για να δίνονται σαφής και ξεκάθαρο λογαριασμό. Όσον αφορά την έκθεση της κυρία Σκοτ Κάτω, υποστηρίζω απόλυτα τα όσα μας είπε. Σα ευχαριστώ. Και τώρα κυρία Ζολή. Madame la Πρόεδρε, συνάδελφοι, ε, κύριε Επίτροπε Μοσκοβισή, το Ευρωκοινοβούλιο κάνει τη δουλειά του. Από το 2009 ψηφίζει φιλόδοξες εκθέσεις όσον αφορά την βελτίωση της ε, φορολόγησης. Όταν μπορεί, το Κοινοβούλιο επιταχύνει τη διαδικασία ώστε να μην καθυστερήσει την πορεία προς καλύτερη νομοθεσία. Όταν ξεσπάει ένα σκάνδαλο, εδώ δημιουργούνται πλειοψηφίες για να ασκηθεί πίεση στους όσους έχουν το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Είναι απαράδεκτο να εμποδίζεται το Κοινοβούλιο να κάνει τη δουλειά του, να στηρίζει την επίγουσα διαφάνεια αναχώρα όσον αφορά τις πολυεθνικές, τα κράτη-μέλη μόλις απαντούν. Και εσείς κύριε αφήνεται να καθυστερεί και να ολισταίνει η συζήτηση. Όταν η Επιτροπή Τάξη ζητά την πρόσβαση σε ουσιαστικά κείμενα για να καταλάβει ποιο άφησε να γίνονται όλα αυτά τα χρόνια όλα αυτά, το δικαίωμά τη ε, περικόπτεται και αγνοείται και τελικά περικόπτεται και παρεμποδίζεται ο δημοκρατικό έλεγχο. Το Κοινοβούλιο δεν είναι το αρχείο το καταγραφής των όσων κάνουν οι άλλοι. Οι ευγενικέ επιστολέ δεν αρκούν. Ο αγώνα για τη δίκαιη φορολογία είναι ένα αγώνα για τη δημοκρατία και θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το καταλάβει αυτό και το μέγεθος, τη σημασία αυτής της ε, υπόθεσης. Ο κύριος Τσάνι Μάρκο. Ευχαριστώ, Το LuxLeaks ε, δεν χρησιμεύσε σε πολλά πράγματα για να αλλάξει ένα επέσχυντο και άδικο σύστημα. Σε μια τέτοια κατάσταση καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην Ευρώπη τα κράτη-μέλη επιδιώκουν ακόμα να εκμεταλλευτούν τους εταίρους τους στην Ευρώπη προς όφελος πάντα των μεγάλων πολυεθνικών που είναι οι μόνες που κερδίζουν πραγματικά αυτή την ε, παράλογη πορεία φορολογικών διευκολύσεων. Ε, το γεγονός αυτό ε, στην ουσία δεν αλλάζει με την κακή συμφωνία στο Συμβούλιο. Όχι μόνο δεν παρέχεται δημοσιοπτήτα στα νομοθετικά κείμενα, στα φορολογικά κείμενα όπως θα έπρεπε, αλλά τα κράτη-μέλη περιορίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μόνο σε διασυνοριακές συμφωνίες, καθυστερώντας την θέση σε ισχύ των κανόνων αυτών, ξεχνώντα ότι έγινε στο παρελθόν. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία βούληση πραγματικά να επιλύσουν το θέμα, προτιμούν να προσελκύουν τι πολυεθνικέ, κάνοντά να πληρώνουν γελία χαμηλά φόρο. Οι μόνοι που, που υφίστανται τι πιέσει είναι οι πολίτε που συνεχώ του ζητούμε περισσότερε θυσίε. Κύριος, η κύριε Καπέλ. Κύριε Καπέλ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Η το θέμα του δαγωνισμού την τελευταία εβδομάδα συζητήθηκε και αναφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι πρώτες δύο υποθέσεις από το σκάνδαλο του λίξ, αυτά τα tax rulings αποτέλεσαν ε, κρατικές επιδοτήσεις, παράνομες. 350 συμφωνίες λοιπόν τέτοιες φορολογικών ελαφρύνσεων ειδικέ ε, συμφωνίες και πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις πήρναν ε, φόρους κάτω από 1% και αυτό οδήγησε σε τεράστιε σημείε, σε τεράστιες απώλειες φορολογικές. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θεωρεί ότι κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνονται 190 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω μετακατάστασης φορολογικών πρακτικών και παρόμοιων φορολογικών πρακτικών. Υπάρχει παρόμοια μελέτη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που αναφέρουν για 50% απώλεια των ατήσεων εσόδων και με πολύ άδικο τρόπο, με στρατηγικές οι οποίες ε, σημαίνουν ότι φορολογούνται κατά 30% οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κάτω από 5% οι μεγάλες. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η σημερινή έκθεση του Μάρκου Βέρμπερ γιατί αποτελεί τον πρώτο συγκεκριμένο βήμα για την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά ζητήματα, σε ό,τι αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις, σε ό,τι αφορά τις φορολογικές συμφωνίες. Εδώ χρειάζεται λοιπόν περισσότερη διαφάνεια σε όλη τη φορολογία προκειμένου να υπάρχει δικαιοσύνη και ανταγωνισμός, να και δίκαιος ανταγωνισμός. Αλλά και στο θέμα της ε, εκθέσεων αναχώρα θα απεριληφθούν τέτοια ζητήματα για κράτη και για ε, επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και θα πρέπει φυσικά να υπάρχει φορολόγηση εκεί που γίνεται το κέρδο για να αναφέρω απλά ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Μάρετιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, εισηγητές που δούλεψαν ε, για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Ενισχύσατε το μήνυμα του Κοινοβουλίου για τη σπουδαιότητα που αποδίδουμε στην διαφάνεια και την σωστή καβολή των φόρων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε ένα σύστημα όπου οι φόροι θα πληρώνονται εκεί που γίνεται η οικονομική δραστηριότητα στην πραγματικότητα. Ε, θέλουμε δηλαδή συστήματα που δεν επιτρέπουν φοροαποφυγή. Χρειαζόμαστε σταθερές, στέρες και προβλέψιμες δομές του φορολογικού, των φορολογικών συστημάτων που θα είναι απλές για τους φορολογητές και για τους φορολογούμενους και θα διευκολυνθούν από την κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις διότι οι αποταμιευτές εισπράττουν ε, εισοδήματα από τις αποταμιεύσεις τους σε μια χώρα ενώ οι αποταμιεύσεις βρίσκονται σε άλλη χώρα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ταυτόχρονα δουλέψαμε πολύ για την ανταλλαγή των φορολογικών πληροφοριών και την συνεργασία μεταξύ χωρών για την κατάργηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Έχουμε τώρα ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τα πρότυπα του ΩΣΑ το πεδίο εφαρμογή της νέας νομοθεσίας είναι ευρύτερο από αυτό της προηγούμενης. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να χάνονται. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να το έχει αυτό υπόψη. Της ευχαριστώ. Βαγιέν, ο επόμενος ομιλητής, πρόεδρε, επίτροπε, συνάδελφοι, όπως συχνά η πραγματικότητα μας προλαβαίνει. Το έδειξε και η Επιτροπή, διότι το ruling που δόθηκε στην ε, Fiat και στο Starbucks ε, στο Λουξεμβούργο και την ε, Ολλανδία αποδείχθηκε ότι ήταν κρυφές και καλυμμένες κρατικές ενισχύσεις. Τα κείμενα που πέρασαν το 11 και το 12 δεν θα επέτρεπαν να γίνουν, εάν εφαρμοζόντουσαν τότε, δεν θα επέτρεπαν να γίνουν αυτές οι παραβιάσεις. Αυτό αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Το κείμενο του Κοινοβουλίου ήταν σαφές, ε, πιο, σαφώς πιο φιλόδοξο από αυτό το Συμβουλίου και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τον κύριο Φέρντα ιδίω και τους κοιόδησε. Προφανώς είναι συμβιβαστικό κείμενο, αλλά θέλω να υπογραμμίσω κάποια σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογής όλες οι αποφάσεις των πολυεθνικών πρέπει να αναλύονται χωρίς εξαίρεση. Είτε είναι εθνικές, είτε διεθνείς και χωρίς προθεσμία. Αλλιώ, γιατί δεν γίνεται αυτό, ποιο θέλουμε να προστατεύσουμε. Δεύτερον, οι κανόνε είναι αποτελεσματικοί αν υπάρχουν κυρώσει, το ξέρουμε. Αυτό ζητά το Κοινοβούλιο, να υπάρχουν κυρώσει αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να συμμετάσχουν ή αν παρέχουν εσφαλμένε ή δεν παρέχουν πληροφορίε. Τρίτον, Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλο τη Επιτροπή στη διαδικασία αυτή. Όλοι ξέρουμε πω δεν μπορεί κάποιο να είναι και δικαστή και διάδικο. Στην πραγματικότητα τα κράτη όμω εδώ αυτό είναι και αυτό θέλει να πετύχει το Συμβούλιο. Τέταρτον, για να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αλλά πραγματική διαφάνεια, όχι μόνο διακοσμητικού χαρακτήρα. Ε, ξέρετε, οι πολλές πληροφορίες σκοτώνουν την ενημέρωση τελικά. Πρέπει να είναι σαφής, προσβάσιμη και κατανοητή ενημέρωση από όλους, όχι μόνο από τους ειδικού. Και τελευταίο σημείο, όλες οι ενεργές, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες πρέπει να έχουν έναν ευρωπαϊκό αριθμό ταυτότητας. Αυτό για να διευκολύνονται η αναζήτησή τους και για να μειωθεί το, το διοικητικό κόστος δεν κερδίζει. Εάν το σύστημα συνεχιστεί δεν χάνει κάποιο κράτος και κερδίζει κάποιο άλλο, αλλά χάνει ένωση συνολικά. Ευχαριστώ κύριε Λούκα. Κύριε Πρόεδρε, εδώ στη συζήτηση αυτή για την έκταση αυτό το θέμα είναι η δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη, προκειμένου κάθε φορολογούμενος να συμβάλλει ό,τι του αντιστοιχεί για την χρηματοδότησή της ε, κοινή ζωής. Και όλοι ξέρουμε από τα έγγραφα του LuxLeaks και από τις ε, έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσίευσε κατά πρώτα πορίσματα την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρχαν μαζικές παραβιάσεις ε, της αρχής αυτής της δικαιοσύνης και διαπίστωσε κρατικές ενισχύσεις μέσω χρηματοπιστωτικών ε, επιχειρήσεων και το, το και τη Starbucks. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι το Συμβούλιο, το Συμβούλιο αποφάσισε τις συνοριακές φορολογικές ελαφρύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην τις καταστήσει προσβάσιμες. Πρόκειται για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για θέματα φορολογικής δικαιοσύνης. Είναι υποχρέωση να καταργηθούν αυτές οι φορολογικές ε, πρακτικές. Ε, θα πρέπει να ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα δεν είναι μόνο να προσαχθούν οι πετοί, Χρειαζόμαστε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις και να πετύχουμε τη δικαιοσύνη που επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λαϊκή Πρόεδρο. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Τόιρερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, τις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του LuxLeaks ένα στοιχείο είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι τα κράτη-μέλη και μια σειρά επιχειρήσεων όντως ε, χρησιμοποίησαν και καμεταλλεύθηκαν συστήματα φοροαποφυγής ύψους ε, δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων και αυτό έχει και καταστροφικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τον ανταγωνισμό που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες ε, πρακτικές και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κατά 25 ε, και παραπάνω ποσοστιαίες μονάδες. Το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής ε, πληροφοριών είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν αποτελεί από μόνο του επαρκή λύση. Μάθαμε για παράδειγμα σε επίσκεψη στην Ελβετία ότι μεταξύ των καντονιών συμφωνήθηκε τη δεκαετία του 50 ένα δίκαιο σύστημα φορολογικό ανταγωνισμού και αυτό συμπεριλαμβάνει και ένα σύστημα φορολογικών ε, πληροφοριών οι οποίες συνταλλάσσονται μεταξύ των μονάδων αυτών. Ζητούμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατεπηγόντως να ρυθμίσει, να φροντίσει να καταργηθούν τα ειδικά καθεστώτα που πρότεινε το Συμβούλιο και αυτό είναι ένα τυρί γεμάτο τρύπε. Ελβετικό, Ολλανδικό, όπω θέλετε, πείτε το. Αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κλείσουν αυτέ οι τρύπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρο. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Βιέγκα. Καταρχήν μια εισαγωγή στα γαλλικά. Ο Γιούνκερ ως ε, υπουργός της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου ε, ε, προέβησε συμφωνίες με εκατοντάδες πολυεθνικές έτσι ώστε να τραβήξει κέρδη προς το Λουξεμβούργο και αυτό σημαίνει κλοπή σε επίπεδο των φορολογικών εσόδων των υπολείπων κρατών μελών. Εμένα διόλου δεν με ενδιαφέρει αν είναι πρόεδρος της Επιτροπής, εφόσον είναι κλέφτης δεν έχει τη δική μου εμπιστοσύνη. Και συνεχίζω στα, γαλλικά, στα πορτογαλικά. Σκάνδαλα φορολογικά, οι ευρωπαϊκές αρχές ε, πρέπει να δεσμευθούν στην καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Ε, να μην είναι μόνο νομοθετικά λόγια, αλλά πραγματικά, πραγματικές θεσμικές υποχρεώσεις. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ελβετία, ο σχετικός ε, κανονισμός περιλαμβάνει διάφορα παραθυράκια. Ε, η Επιτροπή Τάξη έχει παρεμποδίστηκε. Τρεις κυβερνήσεις, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο, αρνήθηκαν την πρόσβαση σε έγγραφα. Όλα αυτά μας οδηγούν στο να αμφισβητήσουμε την πραγματική πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε. Έχετε μπλε κάρτα. Τον κύριο Χέβιτς. Θα απαντήσετε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία σας, ιδιαίτερα το πρώτο τμήμα. Εσείς συμφωνείτε μαζί μου τότε πως αν, εφόσον έχετε αυτά τα αισθήματα για τον κύριο Γιούγκερ και την Επιτροπή του, οτιδήποτε προκύψει από εκεί είναι κάτι που όλοι θα πρέπει να βλέπουμε με μεγάλη προσοχή και καχυποψία και τίποτα που μπορεί να κάνει αυτή η Επιτροπή για αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να μας πείσει, συμφωνείτε με αυτό. Ε, ε, ε, Δεν άκουσα το αρχικό τμήμα τη ερώτησή σα, Θα πρέπει ωστόσο να πω ότι αυτά τα σκάνδαλα αγγίζουν όχι μόνο τον πρόεδρο τη Επιτροπής αλλά και τον πρόεδρο του Eurogroup και τα κύρια κόμματα αυτού του σώματος που στήριξαν όλες τις κυβερνήσεις που άσκησαν για χρόνια και χρόνια ε, ε, αυτή τη διαδικασία, δηλαδή φορολογικές συμφωνίες που είχαν στόχο να ωφελήσουν τις πολυεθνικές και να ε, αποφύγουν την ίση και δίκαιη φορολόγηση. Οπότε αγγίζει όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ίδιο το οικονομικό σύστημα εντός του οποίου τα ιδιωτικά συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών διαρκώς επιβάλλονται στους πολιτικούς. Αυτό είναι το διακύβευμα σήμερα και πρέπει να είναι σαφές. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Οφλίν. Να είμαστε σαφείς. Η ύπαρξη της ίδιας της Ένωσης διευκολύνει τις πολυεθνικές εταιρείε ε, επιθετικά να αποφεύγουν τις ε, δυνητικές φορολογικές υποχρεώσεις τους από, ε, στις ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκούς κανόνες, οι πολυεθνικοί όμιλοι επέλεγαν πού θα καταβάλουν τους φόρους τους ανάλογα με το που ήταν ευνοϊκότερη μεταχείριση. Έτσι, τα μικρότερα κράτη-μέλη της Ένωσης συνήψαν ε, ε, ευνοϊκές συμφωνίες με τις πολυεθνικές και δώσαν την ευκαιρία σε μικροσκοπικά κράτη όπω το Λουξεμβούργο να γίνουν ζάμπλουτα και στις ε, πολυεθνικές να αποφεύγουν τη δίκαιη φορολόγηση στις χώρες που κάνουν τις μεγαλύτερες τους πωλήσει. Οποιαδήποτε λύση λοιπόν με περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη εξουσία στην Κομισιόν δεν θα λειτουργήσει. Η απάντηση είναι τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την κυριαρχία τους στα φορολογικά θέματα για την οικονομική δραστηριότητα εντός των συνόρων τους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίντερ Μάγερ. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την έκθεση για την αυτόματη διαλογή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό βήμα πρόοδου στον τομέα της φορολόγησης. Είναι μια πρωτοβουλία κατά, μεταξύ των πρωτοβουλίων κατά των ΠΕΠΣ που θα διευκολύνει την φορολογία. Το Κοινοβούλιο έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο, αλλά ελπίζω το Κοινοβούλιο να ακούσει τις απόψεις του Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά, γιατί ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση και να παράσχουμε την άποψη και την εμπειρογνωμοσύνη μας. Ελπίζω τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν με τρόπο που θα είναι καλό για το μέλλον τη Ευρώπη και των Ευρωπαίων πολιτών. Να πω επίση ότι πρέπει να αποφύγουμε την ιδέα ότι το καλύτερο είναι πάντα καλό. Αντί να ζητούμε πιο διευρυμένη νομοθεσία θα πρέπει να επιδιώξουμε την καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι το, το περισσότερο δεν είναι πάντα καλύτερο και στον τομέα της καταπολέμησης της φοροαποφυγής. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λούντβιξον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι θετικό το γεγονός ότι μιλάμε για ένα καθολικό πρότυπο ανταλλαγή πληροφοριών και ότι δημιουργείται αυτό το σύστημα και είναι λοιπόν θετικό που θα σε εφαρμογή από το επόμενο έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σημαντικό εργαλείο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αποφυγή της ε, φοροδιαφυγής. Είναι πάρα πολύ λογικό λοιπόν το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, σταδιακή κατάρριξη των εφιστάμενων συστημάτων γιατί δεν θα ήταν λογικό να υπάρχει ένα διπλό σύστημα υποβολή ε, πληροφοριών θα έδινε κάποιες πληροφορίες παραπάνω, αλλά το κόστος, το επιπρόσθετο λόγο της γραφειοκρατίας δεν θα άξιζε τον κόπο. Τα επομενα τρια τρία-τεσσέρα χρόνια είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση της διαφάνειας προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά αυτό το νέο σύστημα. Αυτό όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τα πέντε κράτη που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο καθολικό πρότυπο. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθεί τις εξελίξεις ε, στένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εντοπίσει ενδεχόμενα παραθυράκια. Η υποχρέωση υποβολές εκθέσεων και αναφορών θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο σε στενό κύκλο, αλλά θα πρέπει να χορηγούνται αυτά τα στοιχεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς την ε, κοινή γνώμη. Η μετάβαση αυτό το καθολικό πρότυπο ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το δίνω το λόγο στην κυρία Ρούνα Λέρνεν οι επιχειρήσεις ε, γενικά έχουν την τάση να πληρώνουν φόρο όπως μπορούν και όπου μπορούν. Η περίπτωση των leaks όμως δείχνει ότι δεν συμβαίνει αυτό με όλους. Αν οι πρακτικές αυτές συνεχιστούν, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να χάνουν φορολογικά έσοδα και να μην μπορούν να παράσχουν επαρκή, επαρκείς υπηρεσίε στους πολίτες. Οι φορολογικέ αρχές, κατά την άποψή μου, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικά στοιχεία και οι πολίτες να ξέρουν ποιο πληρώνει τι. Η... Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εντάσεις για το θέμα αυτό. Οι πολίτες ανησυχούν για τα ζητήματα. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία θεωρείται άδικο να προσπαθεί η Πορτογαλία να προσελκύει συνταξιούχος στην Πορτογαλία λέγοντάς τους ότι δεν θα πληρώνουν φόρο εκεί ότι θα περνούν ωραία χειμώνα, θα έχουν ήλιο και θα πληρώνουν και φόρο. Προφανώς η Πορτογαλία είναι μια χώρα με εξαιρετική κοινωνικό επίπεδο ζωής. Αυτό όμως είναι ανησυχητικό. Αυτή η τάση είναι μια ανησυχή τάση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η κυρία Γκουλάρ. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Δυστυχώς η Προεδρία λάμπει δια της απουσίας της. Τέλος πάντων, καλά που είστε κι εσείς εδώ για να συνεχίσετε να ασκείτε πίεση και κατά των ε, διστακτικών κρατών μελών. Δεν πρέπει να βαφκαλιζόμαστε. Το θέμα του ότι προσπαθούμε να βάλουμε λίγο τάξη στο φορολογικό ανταγωνισμό της Ευρώπης, στην Ευρώπη είναι ένα θέμα που, στο οποίο διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Μετά από μία τις αποκαλύψεις για το μέγεθος των φορολογικών αποφάσεων, των ruling στο Λουξεμβούργο, υπάρχει μια απώλεια εμπιστοσύνη. Πολύ καλά λοιπόν ζητάτε περιττέρω ενημέρωση και πληροφορίε. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω ως ε, πρόεδρος της ε, ομάδας για την καταπολέμηση τη ε, της φτώχειας, είναι ότι είδαμε μια έκθεση τον Μάιο που η Επιτροπή λέει ότι η μάχη κατά της φορολογικής ανισότητας περνάει από καλύτερη κατανομή των φορολογικών εσόδων. Χωρίς αυτό δεν γίνεται κάτι. Ο κύριος Ντεμάση. Κυρία Πρόεδρε, η ανταλλαγή αυτή πληροφοριών σε τροδική βάση επί 38 χρόνια δεν λειτουργήσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρησε μέσα στο LuxLeaks. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να πλύνουμε τα... να καθαρίσουμε αυτές τις ε, τα θέματα του παρελθόντος. Οι κεντρικές λοιπόν πληροφορίες για τέτοιες ε, φορολογικές ελαφρύνσεις θα πρέπει να είναι και δημόσιες για να μην υπάρχουν μυστικά. Και στην Επιτροπή είδαμε ότι ήρθε και ο κύριος Γιούγκερ μας είπε τα παραμύθια του χωρίς να μπορέσει να αντισταθεί η πλειοψηφία των βουλευτών. Ακόμα δεν, λάβουμε, δεν λαμβάνουμε λοιπόν επαρκείς πληροφορίες και επαρκή πρόσβαση στα δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρόκειται για ένα μικρό βήμα για το Κοινοβούλιο, αυτό το βήμα που λαμβάνουμε σήμερα, αλλά είναι υπερβολικά μικρό το βήμα αυτό και για το φορολογούμενο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να σταματήσουμε να πούμε, πίεση από πλευρά τη ομάδα μου μέχρι να σταματήσει το φορολογικό αυτό καρτέλ. Ο κύριο Στόλογιαν. În sfârșit, Uniunea Europeană face un pas important pentru a Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτό το σημαντικό βήμα προς την κατευθύνση της ε, πρόληψης ε, της φορολογιαφυγής και φοροποφυγής στα κράτη-μέλη. Με την αυτόματη ανταλλαγή απόψεων, ε, πληροφοριών, κάθε κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση που ένα άλλο κράτος μέλος υπογράψει τέτοιες συμφωνίες που πλήττουν τα συμφέροντα των ε, γειτονικών κρατών. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορες περιστάσεις ζήτησε την εφαρμογή τέτοιων μέτρων και εγώ ίδιος προσωπικά. Αλλά χρειάστηκε ένα διεθνές σκάνδαλο να ξεσπάσει προκειμένου να λάβουμε δράση. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωτοβουλία. Τα παρόλα, Λονόριλη Κάρας. Κύριος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον εισήγητη και όλος ο ιδιαίτερος τον κύριο Φέρμπερ για τις αξιώσεις που θέτει στην έκθεσή του και για τη σημερινή συζήτηση η οποία συνδέεται. Γιατί θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπος Φιστάτσα, καταγγέλει τις, ε, και καταργεί αυτές τις παράνομες φορολογικές πρακτικές και από την άλλη στο LuxLeaks συζητάμε φορολογικές ελαφρύνσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούμε πιο πολύ δικαιοσύνη, πιο πολύ διαφάνεια στην φορολογική πολιτική και τα κράτη-μέλη αρνούνται. Αρνούνται, λέγω, να χορηγήσουν τέτοιε πληροφορίε για τι φορολογικέ αυτέ ελαφρύνσει. Είναι απαράδεκτο. Χρειαζόμαστε πιο πολύ δικαιοσύνη, πιο πολύ διαφάνεια, πιο ίσου όρου. Μία κοινή βάση ανταγωνιστικότητα, μία βάση εκθέσεων χώρα αναχώρα και χορήγηση των φορολογικών αποφάσεων για να υπάρχει πιο πολύ δικαιοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία. La parola onorevole Van Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να μην έχει δικαίωμα να λάβει επίσημες αποφάσεις στο θέμα αυτό, αλλά ζητάμε γενικά έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ανταλλαγή πληροφορίων. Αυτό αποτελεί ένα μήνυμα που δεν μπορεί να το αγνοήσει έτσι απλά το Συμβούλιο. Μόνο δίνοντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κεντρικό ρόλο και πρόσβαση σε βασικέ πληροφορίε για τι φορολογικέ αποφάσει μπορούν να αποφευθούν νέα φορολογικά σκάνδαλα. Και η διστακτικότητα με την οποία τα κράτη-μέλη προσπαθούν να καταπνίξουν αυτό το μέτρο αποτελεί δυσίωνο σημάδι. Γιατί είναι τα ιδρυτικά μέλη εκείνα που διαπιστώσαν ότι η ιστορική αγορά μπορεί να ανθίσει μόνο όταν υπάρχει μια κεντρική υποπτική αρχή, χωρίς ε, να υπάρχουν διαστρεβλωτικοί παράγοντες. Και ακριβώς αυτό ζητάει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί λοιπόν τώρα αυτές οι χρήσιμες πληροφορίες ε, για τις φορολογικές αποφάσεις θα πρέπει να μείνουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μυστήριο αυτό. Και επίσης σκάνδαλο είναι ότι αυτές ε, οι προσπάθειες τάχα για επικυριαρχία κρατική ουσιαστικά στρέφουν τα κράτη-μέλη το ένα κατά του άλλου και τις επιχειρήσεις επίσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμκ. Ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ. Καπούτο. Ούτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλές φορές ε, ζήτησα να ληφθεί υπόψη οι, αρχέ οι αρχές της διαφάνειας ε, σαν βασικές αρχές σε μεταρρυθμίσεις στον εικονικό τομέα. Η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να είναι χρήσιμη μορφή αντιμετώπισης της φοροαποφυγής. Δυστυχώς η ανταλλαγή δεδομένων και η αρχή τη ε, ευθυδικίας δεν είναι πλήρης ακόμα. Ε, δεν, υπάρχουν δεν υπάρχει προληπτική ενημέρωση. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι περιορισμένοι. Τα αποτελέσματα είναι πολύ σοβαρά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την επιβλαβή, ε, τον επιβλαβή φορολογικό ανταγωνισμό. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή για την αναδρομικότητα των ελέγχων των ruling στα 10 χρόνια και τη δυνατότητα εφαρμογή μεγαλύτερη διαφάνεια Είναι αναγκαίο να υπάρξει εμπιστοσύνη και στον τομέα της φορολογίας να αγνοήσουμε μέσω των διοικητικών διαδικασιών που έχουν δεθεί στα κράτη-μέλη Ήρθε ο κύριος Τόμκ. Η κυρία Τόμκ. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτο... ρόλο πρωτοπόρου στην παγκόσμια καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ανταλλάσσουν λίγα στοιχεία για, τα φορολογικά, για τις φορολογικές αποφάσεις. Δεν ενημερώνονται συχνά για rulings που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Εάν υπάρχει υποχρεωτική ενημέρωση θα μειώσει σημαντικά την φοροαποφυγή και την ελκυστικότητα των ευνοϊκότερων φορολογικών συστημάτων. Δεν αρκεί ωστόσο να αντιμετωπίσουμε την ε, φοροαποφυγή. Πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Το ψήφισμα είναι ένα καλό βήμα μπρος, ελπίζω να υπάρξουν και άλλα τέτοια. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μαριά εκτό μικροφώνου. Εκτό μικροφώνου κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν τη σύγχρονη μάστιγα των οικονομιών τη Ευρωζώνη. Πρωταθλητέ στο αντικοινωνικό αυτό σπορ έχουν αναδειχθεί οι πολυεθνικέ επιχειρήσει που μέσα από το σύστημα των ενδοομιλικών συναλλαγών αποφεύγουν την καταβολή φόρων πολλών δις ευρώ. σύμμαχοί τους οι διάφοροι φορολογικοί παράδεισοι και ορισμένα κράτη μέλη της ευρωζώνης που επιδίδονται σε φορολογικό ντάμπινγκ και σε αθέμητες πρακτικές δίνοντας έτσι ζωτικό χώρο στις πολυεθνικές να μην καταβάλουν φόρους πολλών δις ευρώ σε χώρες όπως η ελλάδα εκεί όπου οι πολυεθνικές βγάζουν τα υπερκέρδη τους. το λουξεμβούργο με τα γνωστά luxleaks αλλά και η ολλανδία δίνουν κάλυψη σε γερμανικές και άλλες πολυεθνικές προκειμένου να προαποφύγουν και όλα αυτά τη στιγμή που ο κύριος Ντάισεμπλουμ κουνάει το δάχτυλο στην ελλάδα και απαιτεί νέο φορομπηχτικό ρεσάλτο στις τσάπε του φτωχοποιημένου ελληνικού λαού. επιπλέον κύριε μοσχοβησί η τρόικα στην ελλάδα σφυρίζει αδιάφορα και συγκαλύπτει όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις που αρνούνται να αξιοποιήσουν τη λίστα λαγκάρτ και να φορολογήσουν τους έλληνες ολιγάρχες που έχουν παράνομες καταθέσεις στην ελβετία. γιατί άραγε; Πρόεδρε, ποιον θέλουμε να προστατεύσουμε, αυτό είναι το βασικό θέμα. Τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης ή των πολυεθνικών. Κάποια κρατημέλη, βλέπουμε, λειτουργούν εγωιστικά. Και αυτό είναι εις βάρος των πολιτών προφανώς. Πιστεύω ότι οι προτάσεις είναι θετικές και η ανταλλαγή πληροφοριών υπολογικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που πρέπει να, ε, στο οποίο πρέπει να εμείνουμε για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα μπρος. Έχουμε μια ενιαία αγορά, έχουμε κοινωνόμισμα, το κοινό νόμισμα δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει περάσει σε όλες τις χώρε τη Ευρωπαϊκής αλλά στην πλειοψηφία τους. Το ερώτημα που θέτουμε, πρέπει να θέσουμε ωστόσο, είναι μπορεί να επιβιώσει το κοινό νόμισμα χωρίς κοινή φορολογία. Ο κύριο Σόλτε. Πρόεδρε. Πρόεδρε, Αυξάνεται η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή τα τελευταία χρόνια με μεγάλε ζημιέ για τα κρατημέλη. Χάνονται δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένα προγράμματα του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Προσφάτως ε, είχαμε σαφείς ε, περιπτώσεις ε, φορολογικής κατάχρησης και έλλειψης πληροφοριών. Ε, το κάθε κράτος μέλος θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα στείλει ε, και θα ενημερώσει μάλλον για την τα tax rulings τα οποία εκχωρήχω. Αυτό είναι ό,τι πρέπει για να δημιουργηθούν και άλλα σκάνδαλα. Είναι σωστό λοιπόν να υπάρχει ένα μητρό που θα καταγράφεται ε, όλα αυτά. Μοσχοβή, είναι η παραδοχή όσων κινούνται στην αγορά ότι όσο εμείς συζητάμε εδώ την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή βρίσκουν άλλους δρόμους και τελικά μας προσπερνούν. Γι' αυτό για μένα το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να εφαρμοστεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό σύστημα πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να καταστεί υποχρεωτική στην πράξη πόσο γρήγορα μπορούμε να έχουμε ενιαίο μητρό φορολογία στις επιχειρήσεις πόσο γρήγορα μπορούμε να ξέρουμε πού και ποιοι έχουν καταθέσεις ακίνητη και κινητή περιουσία όχι μόνο μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση αλλά και εκτός αυτής. δεν μπορεί η ευρωπαϊκή ένωση να λειτουργήσει ως νησί και το παράδειγμα της περίφημης λίστας λαγκάρτ στην ελλάδα της λίστας φαλτσιανή που τόσους μύθους καλλιεργεί και τόσα προβλήματα δημιουργεί αυξάνει απλώς το έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες απέναντι στι δυνατότητε μα να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροεπαφυγή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλωσορίζω την συμφωνία που γράφηκε στις 27 Μαΐου 2015 μεταξύ Ένωσης και Ελβετίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα που θα βελτιώσει τη συμμόρφωση και την ενημέρωση. Η Ελβετία είναι ε, κομβικός παίκτη στην ε, αύξηση των προσπάθειών μας να μειώσουμε την φοροποφυγή και φοροδιαφυγή. Πιστεύω ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για λογαριασμούς μεταξύ Ένωση ε, και Ελβετίας που θα ξεκινήσει από το 2018 θα αντιμετωπίσει καταστάσεις όπου ο φορολογούμενος κρύβει, προσπαθεί να κρύψει εισόδημα που, για το οποίο δεν πληρώθηκε φόρος. Επίσης η συμφωνία έχει, θα ενισχύσει και θα επιτρέψει στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών της Ένωσης και της Ελβετίας να εφαρμόσει τη φορολογική νομοθεσία σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Ελπίζω αυτό θα βοηθήσει τις αρχές να εξετάσουν την πιθανολογούμενη παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας και τις πιθανές κυρώσεις αυτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μοσκοβισή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σε κάποιες παρατηρήσεις πολιτικής φύσεως πριν ε, τις διευκρινήσεις. Καταρχήν, συμμερίζομαι απόλυτα την αίσθηση τη συνενετική που διαπίστωσα, όπως την εξέφρασε η κυρία Γκουλάρ, ότι δηλαδή ε, είναι ένα θέμα απόλυτο που αφορά την εμπιστοσύνη. Οι συμπολίτες μας αρχίζουν να αμφισβητούν το δημόσιο λόγο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση αδικίας ε, γιατί καλούνται οι πολίτες να συμβάλλουν ε, ε, στη, στη διάρκεια της κρίσης, ενώ οι πολυεθνικές μπορούν να, εξε, να, εκμεταλλευτούν την τρύπα στην νομοθεσία, το παραθυράκι, για να την κλειτώσουν ε, ή να πληρώσουν λιγότερα εκεί όπου κερδίζουν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αποφασίσουμε από κοινού για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Να προσθέσω ότι είναι και θέμα ε, εμπιστοσύνης αλλά και αποτελεσματικότητας. Γιατί η φοροδιαφυγή δεν έχουμε ακριβή νούμερα γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα έχει κανείς. Ε, μάλιστα θα το δούμε ίσως ε, αφού θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαφάνειας διότι εξορισμού υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία είναι άγνωστα. Πάντως πρόκειται για μια πηγή διόλου αμεληταίων εσόδων για τα δημόσια οικονομία, όπου η δημοσιονομική εξυγίαση είναι απαραίτητη, κυρίως στην Ευρωζώνη, αλλά όχι μόνο σε αυτήν. Εδώ και πολλές μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τοποθετήσει την δίκαιη φορολόγηση και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και φοροαπάτης στις πρώτες της προτεραιότητες. Πιστεύω ότι αν και η κριτική στη δημοκρατική συζήτηση είναι θεμητή, θα πρέπει ωστόσο να φροντίζουμε να μην γινόμαστε λαϊκιστές, να μην κάνουμε να μην ε, ε, δακτυλοδείχνουμε και στιγματίζουμε κάποιους. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, και να καταγγέλουμε την τάδη δίνα προσωπικότητα και η Κομισιόν εδώ ενεργεί και πιστέψτε με με απόλυτα αποφασισμένο τρόπο και καλή την πίστη. Βρίσκομαι εδώ βεβαίω ω Επίτροπο Αρμόδιο για τα φορολογικά θέματα για την θέση μου αυτή, αλλά έχω την απόλυτη εμπιστοσύνη του Προέδρου Γιούνκερ και λευκή επιταγή για να προχωρήσω ε, και μάλιστα χέρι-χέρι ε, συνεργάζομαι με την συνάδελφο Στάγκερ και απαντήσω στην κυρία Ζολή που με χαρά βλέπω εδώ. Ε, μπορώ να σας απαντήσω. Δεν πρέπει να συγχαίομαι τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής με τον αγώνα κατά της Κομισιόν. Πιστεύω πως σε αυτόν τον αγώνα το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν ε, να συνεργαστούν και πρέπει να αγωνιστούν πλάι-πλάι. Εφόσον αναφέρεται τη συνεργασία μεταξύ μας στο πλαίσιο της Επιτροπής Τάξη, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι βρέθηκε συμφωνία με την Επιτροπή Τάξη ώστε οι Ευρωβουλευτές να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που το επιθυμούν. Και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα 89 κείμενα θέσαμε στη διάθεση των Ευρωβουλευτών. 89. Η ε, στάση μας είναι απόλυτα διαφανής και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα κρατημέλη και τις ε, ανάγκες εμπιστευτικότητας ορισμένων στοιχείων από πλευρά των εταιριών. Και έπειτα να πω και δύο λόγια για τα κρατημέλη γιατί άκουσα να δέχονται κριτική εδώ και εγώ ίδιο είπα πριν από λίγο στον κύριο Φέρμπερ σε ποιο βαθμό συμμερίζομαι τη μία ή τη δίνα επικρίσεις του και πόσο πολύ θα ήθελα να είχαμε προχωρήσει περισσότερο σε, σε κάποια σημεία. Όμως ταυτόχρονα τα κρατημέλη τα κράτη-μέλη υπάρχουν και ε, θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία για τη η συμβιβαστική που επαναλαμβάνω είναι καλής ποιότητας είναι ένα σημαντικό μήνυμα ότι και τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να δεσμευτούν για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και γι' αυτό με χαροποιεί. Έχω μια κάποια εμπειρία για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Εδώ ήρθα πρώτη φορά το 1994. Ήμουν μέλος του Συμβουλίου 7 χρόνια, περιλαμβανομένη στις δεκαετίες του 90. Ποτέ δεν είδα ένα φορολογικό κείμενο να εγκρίνεται ομόφωνα μέσα σε 7 μήνες. Με μάλιστα τέτοια καλή διάθεση γιατί αυτό αποδεικνύει ότι αυτό που κάνετε εσείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και εδώ και χρόνια και αυτό που κάνει η Κομισιόν ε, με αποφασιστικό τρόπο οδηγεί στο να κινούνται τα πράγματα. Καταλαβαίνω τις επικρίσεις και ότι δεν έγιναν αρκετά ίσως πράγματα, πάντως προχωράμε. Και η έκθεση που εσείς θα εγκρίνετε υπογραμμίζει ότι όντως πάλι θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Μια επιτυχία θα έχουμε. Και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο επίσης για τη στήριξή του για τα ευρωπαϊκά μέτρα κατά πολέμησης της φοροδιαφυγής, για την προσοχή που αποδίδει στο να προλάβουμε τη χρήση κάποιων τεχνικών για να αποφευθούν ε, αυτά τα μέτρα. Για να ξεφύγει μάλλον κανεί από αυτά τα μέτρα. Τώρα, κάποιες πιο λεπτομερεί απαντήσεις για κάποια ζητήματα που τέθηκαν από τους Ευρωβουλευτές. Καταρχήν το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Αυτό που μου φαίνεται ότι είναι σε αυτή τη φάση η πιο, το πιο σημαντικό σημείο ε, που αναφέρει η έκθεση του Φέρμπερε. Ο εισηγητής θεωρεί πως η οδηγία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις, όλα τα προλογικά έσοδα και όχι μόνο τα έσοδα από αυτά τα, τα rulings, τα διακρατικά, τα διασυνοριακά. Η Κομισιόν είχε από μόνη της περιορίσει, ε, προτείνει μάλλον τον περιορισμό των, της ανταλλαγής πληροφοριών για, ε, στα rulings αυτά. Ε, και το κείμενο του Συμβουλίου αυτή τη στόχο έχει τις συμφωνίες αυτές διασυνοριακές και καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων αποφάσεων. Και γιατί αυτό. Θα έλεγα καταρχήν ότι αν επεκταθούμε σε αποφάσεις που δεν είναι διασυνοριακές θα έχει σαν συνέπεια να αυξηθεί σημαντικά ο φόρτος των των ε, δημοσίων αρχών και ίσως έτσι οι φορολογικές αρχές να μην μπορούσαν να επιστήσουν την προσοχή τους στα κύρια ζητήματα που τις απασχολούν επιπλέον. Ενεργήσαμε επί τη βάση τη νομική που μας προσφέρουν οι συνθήκες που είναι η βάση της εσωτερικής αγοράς. Το να ξέρουμε δηλαδή κατά πόσο τα υπόλοιπα rulings, οι υπόλοιπε ρυθμίσεις ε, καλύπτονται από αυτή τη συνθήκη ε, δεν είναι, το, γνωρίζουμε ακόμα. Πάντως δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι τελείωσε η ιστορία με αυτήν την απόφαση και θεωρώ σκόπιμο το, κύριο, το Ευρωκοινοβούλιο να ξεκινήσει να επιμένει γιατί σε κάποια μεταγενέστερη φάση θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο πάνω σε μια κατάλληλη νομική βάση ώστε να ενισχυθεί η θέση την οποία υποστηρίζει και η Κομισιόν Τώρα, για το θέμα της αναδρομικής ισχύω. Το κείμενο του συμβαστικού του Συμβουλίου προβλέπει μια αναδρομική ισχύ 5 ετών. Είναι πιο σύντομο από τα 10 χρόνια που έχει αρχικά προταθεί. Αλλά θα σας θυμίσω ότι έχουμε ευρύτερο πεδίο εφαρμογή. Καλύπτεται όχι μόνο όλα όσα έχουν ε, ε, δοθεί μέχρι το 2012, αλλά και αυτά ε, που θα έχουν συναυθεί μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου 2016. Προβλέπεται εξαίρεση δε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων ο φοετήσιος κύκλος εργασιών είναι είναι χαμηλός. Ε, έτσι μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη τα επιχειρήματα που μας ε, ε, υποβάλλεται στην τελική πρόταση, ώστε να έχουμε μία πενταετή περίοδο με εξαίρεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι έναν συμπαγή συμβιβασμό. Ο κύριος Μπαγέ με ερώτηση για τον Αφημή. Κομισιόν δεν αποκλεί τη χρήση ενός ευρωπαϊκού αφημί, γιατί, για το, έναν απλούστατο λόγο, γιατί τέτοιο νούμερο δεν υπάρχει ακόμα σήμερα, ωστόσο είναι ένα θέμα ε, επί εργάζεται η Κομισιόν για να μπορέσει να καταπολεμήσει τη φοροποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Είναι ένας τρόπος που θεωρώ εγώ σημαντικό, αλλά δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτιαχτεί ένα τέτοιο νούμερο για να αρχίσουμε να προχωρούμε στην ανταλλαγή πληροφοριών για, τις, για τα rulings. Το, το, τέλος, οι κυρώσεις που κάποιοι αναφέρατε και ήταν ήδη θέμα στην πρώτη μου εισήγηση ενώπιον της Επιτροπής Τάξη. Ο μηχανισμός που επελέξαμε είναι ένας μηχανισμός που στόχο έχει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η διαφάνεια στη συμπεριφορά των πολυεθνικών. Και ε, εγώ βάζω ένα στίχημα εδώ και ελπίζω πως θα το κερδίσουμε και νομίζω πως θα το κερδίσουμε. Η διαφάνεια θα έχει ως αντι, αντι, ε, αποτέλεσμα αντίθετα με τον νόμο του Γκρέσαν που όπως ξέρετε ε, κυνηγά το κακό νόμισμα ε, υπέρ του κακού Θα λειτουργήσει λοιπόν υπέρ τεχνικών πρόβλεψης της θέσης των επιχειρήσεων που οι ίδιες δεν είναι καταδικαστές γιατί δεν, δεν αποφασίσαμε να απο... απαγορεύσουμε κάτι, αλλά να ε, απο... Ε, επιλέξαμε τη διαφάνεια. Πρόκειται για έναν αγώνα, τον οποίο έκανα σώμα με σώμα με αυτούς που πίστευαν ότι ήταν περιττό κάτι τέτοιο. Η παρουσία της Κομισιόν εξασφαλίζει ένα είδο διτητή, που μπορεί μετά να ξεκινήσει διαδικασίες. Και γι' αυτό το λόγο... Και μάλλον και αυτό ακριβώς είναι ε, το έργο που πρέπει να κάνουμε. να έχουμε τέτοιους μηχανισμούς ώστε να έχουμε και πιο συμπαγείς βάσεις με τη νέα οδηγία που πιστεύω θα εγκριθεί μετά από την πρόταση της Κομισιόν, τη Συμφωνία του Συμβουλίου και τη δική σας, της δικής σας έκθεσης. Ο αγώνας για τη διαφάνεια δεν πρόκειται να πάψει. Μιλώ εγώ εδώ για την επανάσταση της διαφάνειας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω για τη δική μας πολιτική αποφασιστικότητα. Ξέρετε, ε, για την πολιτική φυσικότητα της Κομισιόν και τη δική μου προσωπικά. Και το λέω και όσα είπα στην εισήγησή μου, ότι δηλαδή η Κομισιόν θέλει να βάλει το άξιση CCTB που θα περιλαμβάνει την εξυγίανση που είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις για τους λόγους που αναφέραμε που αφορούν την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Επαναλαμβάνω ότι ε, η Επιτροπή θέλει να δείξει ε, ποια ε, μπορεί να είναι τα ωφέλη μιας αποτελεσματικής φορολόγησης. Είμαστε σε μια κατάσταση που μια πολυεθνική εταιρεία δεν πληρώνει καθόλου φόρους ή ελάχιστος εν εκεί όπου βγάζει τα κέρδη της. Και εκεί είναι θέμα εμπιστοσύνη και πρέπει να λυθεί το θέμα. Τέλο, η Επιτροπή εργάζεται στις, για τι εκθέσει αναχώρα, αναφορέ αναχώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο θα ήθελα να μα έχει λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη και να έχει λίγο μεγαλύτερη υπομονή. Με τον συνάδελφο Τζόναθαν Χίλ προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κάτι που καταρχήν ξεκίνησε με μια διαβούλευση. Και στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί σε μια αξιολόγηση όχι για να ξεφύγουμε από το θέμα, αλλά για να δούμε υπό ποιε συνθήκες η αναφορά ανά χώρα μπορεί να συνδυάσει τη διαφάνεια και την οικονομική αποτελεσματικότητα χωρίς να επιβαρύνει τις επενδύσεις των επιχειρήσεων, που είναι απαραίτητες για την απασχόληση. Εγώ προσωπικά εξέφρασα σαφή πολιτική προτίμηση, δηλαδή πρόσβαση του κοινού, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την οικονομική πραγματικότητα. Οπότε έχουμε ε, τις εξή εναλλακτικέ. Είτε ακολουθούμε αυτό που λέει ο που προτείνει, σα θυμίζω, να μείνουμε στις ανταλλαγέ ανάμεσα στις διοικήσεις ή αντίθετα να προχωρήσουμε περισσότερο και παραλαμβάνω ότι είναι δική μου προσωπική προτίμηση με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ε, τιμωρεί, δεν επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και κύριοι βουλευτές σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τους σκιώδη εισηγητές για την εργασία τους. Πιστεύω ότι πέρα από τις διαφορές μας όλοι είμαστε ενωμένοι και θεωρούμε ότι υπάρχει μια νέα πολιτική βούληση που επιτρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ και πιο γρήγορα. Και εσείς εκεί συμβάλλατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ομιλία για το φορολογικό, τα φορολογικά ζητήματα, το οποίο ξεπερνάει φυσικά ε, τα θέματα τα οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε σήμερα και αύριο. Αλλά σας ευχαριστώ. Και λυπάμαι ιδιαίτερα που δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου εδώ, γιατί πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ως κριτική σήμερα δεν απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά προς τα δεξιά σας, τα δεξιά μου, προς το Συμβούλιο και Λάμπιμ για τις απουσίες του. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει το Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί σοβαρό εταίρο και σε φορολογικά ζητήματα. Προσπάθησα λοιπόν να ε, ξεκαθαρίσω την, το ρόλο μας αυτόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και τους συζητητές για την καλή συνεργασία, γιατί σε μέσα, πολύ, σε, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να επεξεργαστούμε και ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Και ελπίζω αύριο να στέλνουμε ένα σαφές ηχηρό μήνυμα προς το Συμβούλιο με μια ισχυρή πλειοψηφία. Αυτό το Συμβούλιο το στέλνουμε προς το Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, όχι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή έκανε ό,τι της αναλογούσε στα θέματα tax rulings. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί το Συμβούλιο αυτά που προτείνουμε. Γιατί ως Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι αυτά που προτείνουμε θα προωθήσουν τη διαφάνεια και την δικαιοσύνη στα φορολογικά ζητήματα και αυτό θα έπρεπε να θεωρούν ε, προς όφελός τους τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Σίμων. Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ τον ε, εισηγητή ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να παραβρεθεί. Εκπροσωπώ την, την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω κάποια λόγια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Φέρμπερ καταρχά, Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστούμε στα θέματα αυτά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για πολλά από αυτά που έχουμε πετύχει, αλλά παράλληλα θέλουμε να βάλουμε και το δάχτυλο στην πληγή εκεί όπου θεωρούμε ότι δεν φτάνει η δράση μα. Και σε ό,τι αφορά τη δράση τη Ειδική Επιτροπή, θα έπρεπε να σα πω ότι σήμερα έλαβα μία πληροφορία η οποία μου προκαλεί κάπω σύγχυση και θα επηρεάσει τις ε, εργασίες μας. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ταχθήκε υπέρ της διαφάνειας και υπέρ της διάθεσης στο, Συμβουλίο, στο Κοινοβούλιο των εγγράφων που ζητήσαμε. Σήμερα λοιπόν έμαθα ότι τα ίδια έγγραφα, τα ίδια τεκμήρια τα οποία μας διατίθονται υπό συγκεκριμένου όρους ε, δημοσιεύθηκαν για μελέτες ε, και μάλλον κοινοποιήθηκαν, δημοσιεύθηκαν, κοινοποιήθηκαν σε ερευνητικά κέντρα με το κανονικό καθεστώς πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Αν αυτό ισχύει, υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω ότι σήμερα δεν θα μπορέσετε ασφαλώς να απαντήσετε εκτεταμένα στο θέμα αυτό, αλλά θα σας το θέσω και γραπτά το θέμα αυτό, γιατί είναι δύσκολο βάσει των εγγράφων που έχουμε στη διάθεσή μας να εργαστούμε ε, επικοδομητικά. Αλλά αν υπάρχουν και χορηγούνται τα έγγραφα αυτά ήδη, θα επιμείνουμε να έχουμε ίση αντιμετώπιση όπως και τρίτη. Νομίζω ότι αυτό το απαιτεί η αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου. Σκοτ Κλείνοντας τη συζήτηση αυτή, Πρόεδρε, να σημειώσω ότι απέδειξε σαφώς πόσο κοινή συμφωνία υπήρξε μεταξύ των συναδέλφων. Πολλά θέματα συμφωνούμε απόλυτα, πολλά θέματα συμφωνούμε απόλυτα. Υπήρξε μεγάλη υποστήριξη σκιώδησή της. Επίσης, το Κοινοβούλιο ανέλαβε δράση στον τομέα αυτό εν λόγω και του, της δημόσιας κατακραυγής αλλά και γιατί στην Επιτροπή Τάξ πήραμε περισσότερες πληροφορίες και αυτό είναι από τα μεγάλα επιτεύγματα. Για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας χρειαζόμαστε πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία. Και χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για διάθεση περιττέρου κειμένων αλλά ε, το να έχουμε κείμενα σε μια αίθουσα, ένα αναγνωστήριο δεν αρκεί. Δεν μοιάζει διαφάνεια να έχουμε και καλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση. Επίσης, πρέπει να πάυσει η επίθεση κατά των πληροφοριοδοτών που βρουν προς όφελος του δημόσιου συμφέροντας. Εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότιμη αντιμετώπιση ε, φορολογικά των επιχειρήσεων που των μεγάλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν να μειώσουν το φορολογικό τους βάρος εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμπερ και να συμφωνήσω μαζί του ζητώντας τη συμμετοχή των κρατών μελών. Υποστηρίζουμε την, ε, θέλουμε την υποστήριξη της Κομισιόν αλλά και των κρατών μελών. το τέλος της φοροποφυγής είναι πήγουσα προτεραιότητα για όλους μας και για μας και τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση ούτε Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο.